Θα ξεκινήσουμε από το σημείο 8 τοποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για τη στήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου. Έχουμε ήδη συζητήσει την έκθεση αυτή, μπορούμε να περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία νομίζω. Ξεκινάμε με την 8, μετά θα συνεχίσουμε με την 9, μετά θα μιλήσουμε για την άμεση στήριξη και μετά για τα αντιβιωτικά. Λοιπόν έχουμε τρεις ψηφοφορίες, θα τις ξεκινήσουμε τώρα για να μπορέσουμε μετά να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Λοιπόν δεν βλέπω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την πρόταση που σας έκανα. Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Μιλάμε για την ευθυγράμμιση τώρα με τη συνθήκη. Είστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαρίθμε νέα. Α, όχι, για μια στιγμή, μια στιγμή λέει ο Πρόεδρος. Πρώτα θα πρέπει να ψηφίσουμε την τέσσερα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ψηφίζουμε λοιπόν την τέσσερα. Πέρα της ψηφοφορίας για την τροπολογία της Επιτροπής Ανάπτυξης απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα την 9, ταραμπέλα. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, η 9 γίνεται δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την υπαριθμητρία 3 του εισηγητή. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφθηκε η τρία. Ψηφίζουμε την δέκα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας δεκτή. Η 11 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε τώρα την 4. 4 ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Περνάμε στην 5. Πάντα του εισηγητή. Ψηφίζουμε την 5. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Περνάμε στην 12. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Η 6. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 6 του εισηγητή. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. Φτάνουμε στην 13, Λαβία. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 13. Τέλος. Δεκτή. Και τώρα φτάνουμε σε ομαδική ψήφο, στο σημαντικότερο ίσως κομμάτι αν θέλετε, τις τροπολογίες 7, 8, 1 και 2. Ψηφίζουμε. Τέλος, ομόφωνα δεκτή η πρόταση ή οι τροπολογίες αυτές δεκτές. Έχουμε άλλες τρεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στις αιτιολογικές σκέψεις 13. Ψηφίζουμε την 1. Τέλος. Απερίφθη οι δύο ψηφίζουμε τέλος απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα την 3. Τέλος. Ψηφίσατε όλοι. Απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της τροπολογημένης πρότασης, νομοθετικής πρότασης. Ψηφίζουμε. Τέλος. Τώρα θα ψηφίσουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Τέλος. Ε, Και τέλος, <clears throat> τελική απόφαση. για τις διαπραγματεύσεις, διορθώνει ο Πρόεδρος. Τελική ψήφος για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ψηφίζουμε. Τέλος. Bene, a larga maggioranza Εγκρίναμε λοιπόν την πρώτη έκθεση. Ευχαριστώ τον εισηγητή, λέει ο πρόεδρος. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ψήφο, ψηφοφορία μάλλον, τροποποίηση του κανονισμού 73 του 2009 κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους διοργούς. Και αυτό είναι ένα κείμενο που αφορά την ευθυγράμμιση τη λεγόμενη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία παριθμών 4. Ψήφισαν όλοι, πέραση τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την 29. Τροπολογία 29. Πέρας εγκρίνεται. Άρχεται ψηφοφορία για την 30. 30. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 5 του εισηγητή. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 31. Ψήφισαν όλοι για την 31. Καλώς, πέραση ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 7. 7. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα την 32. Άρχεται η ψηφοφορία για την 32. Πέραση της πληροφορίας εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην 34. 34. Άρχεται η ψηφοφορία για την 34. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε την 35. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία, εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 36. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ψηφίσουμε τώρα την 37. Πέρασες ψηφοφορίας για την 37. Απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 38. Πέρασες ψηφοφορίας ψηφοφορία για την 38. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 39. Ψηφίζουμε για την 39. Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορία για την 39. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 9. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 10. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 10. Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 11. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία υπαριθμών 12. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 12. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Άρχεται τώρα η ψηφοφορία για τη 14. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τροπολογία υπαριθμών 40. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη 40. πέρα τη 40 απορρίφθηκε. επειδή απορρίφθηκε η τροπολογία υπαριθμό 40, υπάρχει μια πρόταση προφορικής τροπολογίας από τον συνάδελφο Λενίτσκα. Θέλετε να πείτε κάτι ή υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι αντίθετος ε, στην ε, προφορική τροπολογία. Ωραία. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μου η πρόταση είναι η εξής στον ορισμό της κληρονομιάς, επειδή αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε εθνικά νομοθετικά συστήματα, ο ορισμός να παραμείνει στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Να γίνει μια επαναδιατύπωση με τον εξή τρόπο δηλαδή. Οι διατάξεις που αφορούν τον ορισμό της κληρονομιάς της εθνικής νομοθεσίας θα πρέπει να παραμείνουν όλα αυτά στο άρθρο 43. Καλώς. Αν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, να έχει ενστάσεις για αυτή την προφορική τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τροπολογία υπαριθμό 41. Άρχεται η ψηφοφορία για την 41. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία υπαριθμό 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για τη 42. Πέρασε τη ψηφοφορία για τη 42. Απορρίπτεται. 43. Άρχεται η ψηφοφορία για την υπαριθμό 43. Πέρασε τη ψηφοφορία για τη 43. Έγκρινεται. 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία υπαριθμών 16. Πέρασε τη ψηφοφορία για τη 16. Απορρίπτεται νομίζω. 44. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 44. Μενταμέντο 44. Τροπολογία 44. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 17 του εισηγητή. 17. Ψήφισαν όλοι. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται 17. Τροπολογία υπαριθμό 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία για τη 18. Τροπολογία 18. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία για την 20. Ψήφισαν όλοι. Ευχαριστώ. Καλώς πέρασε ψηφοφορίες για την 20. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 22 και 23 που είναι πανομοιότυπη. 22 και 23 μαζί άρχεται η ψηφοφορία για τις 22 και 23 από κοινού. Εγκρίνονται. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 45. 45. 45. Ψήφισαν όλοι τη 45. Πέρασε ψηφοφορία για τη 45. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 46. Άρχεται η ψηφοφορία για την υπαριθμό 46. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Άρχεται τώρα η ψηφοφορία για τη 47. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 47. Πέρα στις ψηφοφορίες για τη 47. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα unblock Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία για τις 24, 25, 26, 1, 2 και 3. Άρχεται η ψηφοφορία για την unblock τροπολογίες. Πέρασε η ψηφοφορία, συγκρίθηκαν ε, ψήφισαν όλοι εγκρίνονται. Και ψηφίζουμε τώρα την 48. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 48. Πέρασε τη ψηφοφορία για τη 48 απορρίπτεται. Περνάμε στην 27, τροπολογία 27, άρχεται η ψηφοφορία για την 27, πέραση της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε τώρα για την νομοθετική πρόταση ως τροποποιήθηκε. Τελική ψηφοφορία για την νομοθετική τρόπο, πρόταση ως τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι. Καλώς εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Καλώς, εγκρίθηκε. Και τέλος ψηφίζουμε για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Εν της έγκρισης της ε, συμφωνίας πρώτης ανάγνωσης. Τελική ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι. Καλώς. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. η δεύτερη τροποποίηση του κανονισμού. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή, λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε τώρα στο σημείο παριθμών 10, η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Θέλει να λάβει το λόγο ο Αντιπρόεδρος. Παρακαλώ. Ο λόγος στον Αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Γιατί ήταν πραγματικά ε, εύκολο το έργο που μου αναθέσατε. Ήταν πάρα πολύ εύκολο στο σημείο αυτό να βρούμε συμφωνία σε 35 από τα 38 ζητήματα. Τώρα απομένουν λίγα ανοιχτά θέματα στα οποία δεν συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά ανεξάρτητα από το αν θα εγκριθούν ή όχι τα θέματα αυτά, δεν πρόκειται να τροποποιήσουν ουσιαστικά το κείμενο. Η πρόταση 39 αφορά τους κτηνιάτρους. Θεωρώ ότι αυτά που προβλέπονται δεν είναι απόλυτα δίκαια και μάλλον θα οδηγήσουν σε δυσκολίες. Νομίζω ότι θα δυσκολέψουν περαιτέρω την εργασία των ε, κτηνιάτρων. Για την 50 δεν συμφωνούμε καθόλου. Υπάρχει ένα λόμπι με λανθασμένα στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν ε, και κάποια στατιστικά στοιχεία από τη Δανία, όπου κάποιες οργανώσεις σε ό,τι αφορά τα αντιβιωτικά. Καταδεικνύουν μάλλον ε, οι έρευνες αυτές ότι έχει αυξηθεί η χρήση αντιβιωτικών στα ζώα. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες ε, αναφορές. Εγώ πάντως προτείνω προσωπικά να υπερψηφίσουμε την πρόταση αυτή. Η διατύπωση τελικά είναι όσο πιο αδύναμη γίνεται. Δεν προβλέπονται επιταγές, διατάξεις, προδιαγραφές. Και τελευταίο στοιχείο για την προστασία των ζώων, την ε, υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία. Όπως και αν το αναφέρουμε, το θέμα δεν είναι αυτό γιατί ξέρουμε ότι η σχέση ψυχικής και σωματικής υγείας είναι άρρηκτη το well-being τώρα στα αγγλικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα, για τα θηλαστικά και για όλα τα ζώα. Όπως αναφέρει ο κύριος Δεκάστρο στην 55 τροπολογία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Πόλσεν και αν συμφωνείτε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έτοιμοι. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 30. Iniziamo sul 30. 30. Ψήφισαν όλοι, πέρασε τις ψηφοφορίες για τη 30, εγκρίθηκε. Ομόφωνα. 31. Τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία για την 31. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία για την 31. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία για την 32. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία για την 33. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία εγκρίθηκε. Οι 34 και 35 από κοινού. Ψηφίζουμε λοιπόν τις 34 και 35 μαζί. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία ψηφοφορίας εγκρίθηκαν. Τροπολογία 36. Άρχεται η ψηφοφορία για την 36. πέρασε ψηφοφορία ψηφοφορίας για την 36. Απορρίπτω. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο, κύριο, Χάουσλινγκ. 37 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 37. Πέραση ψηφοφορία ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 38. Άρχεται η ψηφοφορία για την 38 εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε την 39. Άρχεται η ψηφοφορία για την 39. Πέρασε τις ψηφοφορίες για την 39. Εγκρίθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 40. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 40. Πέρασε της ψηφοφορίας για τη 40. Εγκρίθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 41. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στη 43. Άρχεται η ψηφοφορία τη 43 Πέρασε της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 44. Άρχεται τη ψηφοφορία για τη 44. Πέρασε τη ψηφοφορία για τη 44. Εγκρίθηκε. 45. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 45. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. για τη 46 έως 49 μπλοκ. 46, 47, 48 και 49 μπλοκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Άλλο, άρα θα τις πάμε μία-μία. Ψηφίζουμε μόνο τη 46. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 46. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε τη 47. Είπαμε μία-μία θα τις κάνουμε. 47. Πέρασε της ψηφοφορίας για τη 47. Απορρίφθηκε. εγρίνεται. Όταν έχουμε ίσες ψήφους, λέει ο πρόεδρος, ε, σημαίνει ότι εγκρίνεται. 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 48. Εγκρίνεται. 49. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 49. Chiusa su 49. Πέρασε τι προφορέ για τι 49. Εγκρίθηκε. Ο κύριος Ταραμπέλα. Παρακαλώ. Ο κύριος Ταραμπέλα έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να μας εξηγήσετε γιατί γίνεται δεκτή η ε, πρόταση όταν έχουμε ίση, ο αριθμό ψήφων. Όταν πρόκειται για παράγραφο, ναι. Εδώ όμω έχουμε τροπολογία, τροπολογία υπαριθμό 47, ίσως αριθμό ψήφων σημαίνει ότι απορρίπτεται. Πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία για να γίνει αποδεκτή. Έτσι νομίζω. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ευχαριστώ Μάρκ. Η γραμματεία λέει ότι έχεις δίκιο. Επομένως η τροπολογία περθμό 47 απορρίπτεται. Ευχαριστώ Μάρκ. Συνεχίζουμε τώρα. Τροπολογία υπαριθμών 50. Άρχεται η ψηφοφορία για την 50. Πέρασε τις ψηφοφορίες για την 50. Ψηφίζουμε για την 50, συγγνώμη, είναι ακόμα ανοιχτή η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι για την τροπολογία 50. Καλώς, πέρασε τις ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 51. Άρχεται η ψηφοφορία για την 51. Ψήφισαν όλοι. Καλώς. Η 51 εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 53. 53. Ψήφισαν όλοι για την 53. Καλώς. Εγκρίνεται η 53. Ψηφίζουμε την τροπολογία 54. Άρχεται η ψηφοφορία για την 54. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λάθος λέει ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμός 54. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία τώρα. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 55. Άρχεται η ψηφοφορία για την 55. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται η 55. Τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 1. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 2. Πέραση η ψηφοφορία για τη 2 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία υπαριθμών 3. Άρχεται η ψηφοφορία για την 3. Πέρασε τις ψηφοφορία για την 3. Απορρίπτεται νομίζω. Ισοψηφία έχουμε. Ο κύριος Λεφόλ λέει ότι υπάρχει μία ψήφος ακόμα, πρέπει να ξαναψηφίσουμε, γιατί ε, δεν ε, πατήθηκε το κουμπί του κύριου Ταραμπέλα. Ξαναψηφίσουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπεριθμών 3. Πόλσεν, Σαλτεμό, Εμποβέ και άλλου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 4. Γέγκλε Ματιέ. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 4 πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα για την 5. Πέρας της ψηφοφορίας για το πρώτο τμήμα εγκρίνεται και περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα και πάλι για την τροπολογία υπαριθμό 4, δεύτερο τμήμα. Ψήφισαν όλοι, εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε με τις αιτιολογικές σκέψεις. Sul 5. Τροπολογία 5. Πέρασε η ψηφοφορία για την 5, εγκρίθηκε. Θέλετε να ψηφίσουμε unblock. Να ψηφίσουμε unblock τις 6, 7, 8, 9, 10 και 11. Συμφωνείτε. Τις ψηφίζουμε όλες μαζί. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. Ομόφωνα σχεδόν. Τη 12 τώρα. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση τη ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. 13. Πέρασε τις για τη 13. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 15. Πέραση τη ψηφοφορία. απορρίπτεται. 16. Πέρας τις ψηφοφορίες για τη 16 ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. Η 16 απορρίπτεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 17. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 18. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες για τη 18. Απορρίφθηκε. 19. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 19. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20. Άρχεται η ψηφοφορία για την 20. εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία για την 21. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 22. Άρχεται η ψηφοφορία για την 22. Πέρασε η ψηφοφορίας για την 22. Άρχεται την ψηφοφορία για την 23. Πέρασε τη πληροφορία για την 23. Εγκρίνεται. Έχουμε τώρα μια προφορική τροπολογία. Κυρία Πόλσεν, θέλει το λόγο για την προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να διευκρινίσω ότι η χορήγηση αντιβιωτικών σε προληπτικό επίπεδο ή η χορήγηση αντιβιωτικών για την ανάπτυξη την ταχύτερη των ζώων είναι κάτι το απαγορευμένο στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς η απαγόρευση αυτή δεν ελέγχεται εάν πράγματι εφαρμόζεται. Συνεπώς εφόσον δεν υπάρχει έλεγχος οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση είναι άχρηστη. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, ωραία είναι όλοι υπέρ. Ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 25. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία για την 25. πέρασε της ψηφοφορίας. 26. Άρχεται η ψηφοφορία για την 26. Εγκρίνεται. πέρασε της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία για την 27. Άρχεται η ψηφοφορία για την 27, είπαμε. πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 28. Πέρασε η ψηφοφορίας για την 28. 29. Άρχεται η ψηφοφορία για την 29, πέρασε ψηφοφορία για την 29, εγκρίνεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Καλώς με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστούμε κυρία Πόλσεν. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή έχει ήδη έρθει ο Επίτροπος Τζον Ντάλι, θα κάνουμε ένα μικρό, μια μικρή τροποποίηση. Ο Μάρτιν, συγγνώμη, ο Επίτροπος Ντάλι ήρθε, επομένως θα τον αφήσουμε να περάσει και να ακούσουμε τα του προγράμματος του χαρτοφυλακίου του.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 Bene, se siamo pronti Ξεκινάμε για μια ακόμη φορά. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Τζον Ντάλι. Ο Επίτροπος Τζον Ντάλι είναι υπεύθυνος για θέματα υγείας και για θέματα καταναλωτών θα του ζητήσουμε να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας του για το 2012 στα πλαίσια ενός διαλόγου για ισχυρότερη συνεργασία μάλλον ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία του εδώ. Μετά από την παρουσίασή σας, συνάδελφοι μπορούν να θέσουν ερωτήσεις και θα ακολουθήσει συζήτηση. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, καλημέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας ένα χρόνο μετά από την ανάληψη της εντολής μου και ένα χρόνο μετά από τότε που σας είχα απευθύνει για πρώτη φορά το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερως τις προτάσεις σας και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου γενικότερα και προσβλέπω σε μία περαιτέρω καρποφόρο και επιτυχή συνεργασία. Με την ευκαιρία αυτή θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα του προγράμματός μας για τον επόμενο χρόνο και να αναφερθώ και σε κάποια τρέχοντα θέματα χωρίς να προσπαθήσω να καλύψω όλα τα θέματα. Είναι σαφές ότι θα υπάρξουν ε, πολλές διαφορετικές ε, ερωτήσεις οι οποίες θα συμπληρώσουν τις δικές σας ανησυχίες. Σχετικά με την υγεία των ζώων στις κτηνοτροφικές δραστηριότητες βασική αρχή είναι η πρόληψη. Όλοι γνωρίζουμε τις πολύ αρνητικές πλευρές που έχουν ζωνώσει στα, στις οικονομικές εκμεταλλ... στα οικονομικά των κτηνοτροφικών μονάδων. Απαιτείται να υπάρχει μία πιο αηφόρος και ε, κερδοφόρος ταυτόχρονα ε, ακτινοτροφική διαδικασία πρέπει να καταπολεμούνται ε, οι ασθένειες των ζώων όπου αυτές εμφανίζονται και γι' αυτό νομίζω ότι η τελική μας πρόταση να γίνει δεκτή φέτος ή μάλλον όχι φέτος, του χρόνου θα γίνει δεκτή η η το νέο σύνολο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διευκρινίζει τις ευθύνες των κτηνοτρόφων, των επιχειρήσεων, ε, των κρατικών αρχών και των μέτρων πρόληψης των ζωονόσων, της μείωσης των κινδύνων από τις ζωονόσους και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι νέες προτάσεις μας θα μας επιτρέψουν να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες όπως οι λεγόμενες αναδιόμενες ζωνώσει και να λάβουμε υπόψη μας τα νέα μέσα που μας δίνει η τεχνολογία όπως νέες μορφές εμβολιασμού ή νέα συστήματα ανείχνευσης και ελέγχου των ζώων. Τέλος, ο νέος νόμος θα μας δώσει νέα θεμέλια, περαιτέρω θα έλεγα καταγραφής των προτεραιοτήτων από το 2012 και μετά. Οι προτάσεις αυτές θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε τα κοινοτικά μέσα και τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι νέες αυτές νομικές ε, ρυθμίσεις θα συνοδευθούν από τροπολόγηση των ε, κανονισμών για τους ελέγχους της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και της υγείας ε, των ζώων. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν σαν στόχο να απλουστεύσουν και να καταστήσουν πιο αποδοτικό το παρόν σύστημα και ταυτόχρονα πιο ενιαίο στο σύνολο της Ένωσης. Υπάρχει δυνατότητα επίσης περαιτέρω βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών διαδικασιών μέσω τελών που θα ζητούνται από τις επιχειρήσεις. Θα υπάρξουν λοιπόν οι απαιτούμενες νομικές αλλαγές για την αναθεώρηση και ε, ε, των μέτρων στον τομέα της κτηνοτροφίας και της γεωργίας επίσης και της πορείας ταυτόχρονα. Απαιτείται ε, πριν από οτιδήποτε άλλο να περάσουμε σε εξυγχρονισμό των μορφών ελέγχου. Θα πρέπει οι έλεγχοι αυτοί να χρησιμοποιούν νέες εναρμονισμένες μορφές ενιαίες για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να ξεπεράσουμε την πολυδιάσπαση που χαρακτηρίζει τους ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο για το σύνολο του ευρωπαϊκού εδάφους, μια τέτοια συνολική αντίληψη περιλαμβάνει ε, κτηνο, κτηνιατρικές, ε, τελωνιακές, ε, κτηνιατρικούς τελωνιακούς ελέγχους, Μέχρι τώρα οι κανόνες που είχαμε ήταν σχετικά αποτελεσματικοί, αλλά ήσαν πολύ περίπλοκοι και θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία σε άλλους τομείς. Ε, πρέπει να υπάρξει αύξηση των λεγόμενων φυσικών ελέγχων, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα τεχνολογικά δεδομένα που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας και τις δυνατότητες συλλογής και επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων έτσι ώστε ε, τα ελεγκτικά μας μέσα να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά και οι έλεγχοι στα εξωτερικά μας σύνορα ε, να αρμόζουν κάθε φορά στα προφίλ επικίνδυνοτητας ζώων, φυτών ή ζωοτροφών. Νομίζω ότι αυτή η συνολική αντίληψη θα ενισχύσει τη συνεκτικότητα, αποτελεσματικότητα και εναρμόνιση του ελεγκτικού μηχανισμού συνολικά προς όφελος και των καταναλωτών αλλά και των διοικητικών μηχανισμών. Το πρόγραμμα εργασίας για το 2012 προβλέπει ρυθμίσεις επίσης και θέμα για ρυθμίσεις για την υγεία των φυτών. Καταπολέμηση επίσης βλαβερών οργανισμών από τρίτες χώρες. Είναι βασικό να προστατεύσουμε την γεωργία, την δασοκομεία από ε, ξένες εισαγόμενες ασθένειες και ζυζάνια. Η παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει την εισβολή θα έλεγα τέτοιων ουσιών και ζυζανίων και ακριβώς το ελεύθερο εμπόριο μας καθιστά πιο ευάλωτους. Μια αξιολόγηση του καθεστώτος υγείας των φυτών θα οδηγήσει σε προληπτικές δράσεις. Η έλλειψη πόρων η οποία παρατηρήθηκε περιορίζει την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος ελέγχου και οδηγεί σε εκ των υψηλά κόστη. Πρέπει να αντιμετωπιστεί λοιπόν το θέμα των περισσότερων πιστώσεων στα πλαίσια του πολιετούς προγράμματος 2014-2020. Η πρόληψη είναι η καλύτερη συνταγή και είναι φυσικά και ευθυνότερη μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει και για τα φυτά και ε, για τα ζώα. Να αναφέρω επίσης ότι τα πολλαπλαστικά μέσα και οι ρυθμίσεις οι νομικές γύρω από τα πολλαπλασιαστικά μέσα, σπόροι κτλ. θα γίνουν αντικείμενο περαιτέρω ρυθμίσεων. Να έλθω τώρα στο θέμα της ευημερία των ζώων. Θα παρουσιάσω μια έκθεση το φθινόπωρο για τη μεταφορά των ζώων. Βασικός στόχος θα είναι να καθοριστούν οι κανόνες με ξεκάθαρο τρόπο για την εφαρμογή της οδηγίας για τη μεταφορά των ζώων και να εντοπίσουμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους καταπολέμησης των προβλημάτων που ανεφάνισαν. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια νέα στρατηγική για την ευημερία των ζώων πριν το τέλος του ενεστώτος έτους, τον προηγούμενο Μάιο. Το Κοινοβούλιο σας υιοθέτησε την έκθεση Πόλσον σχετικά με τις πολιτικές που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα και ζητούσε να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική. Το Κοινοβούλιο ζητούσε ιδιαίτερο την υιοθέτηση ενός γενικότερου νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευημερία του ζώου και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Αναφοράς. Οι προτάσει του Κοινοβουλίου είναι αντικείμενο σοβαρής εξέτασης από πλευρά μας. Περαιτέρω δράσεις, εφαρμογή και εναρμόνισης είναι προαπαιτούμενες. Η επιβολή των κανόνων για την ευημερία των ζώων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει οι μέθοδοι που ακολουθούμε να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Να τελευταία λοιπόν, ε, την κάλυψη συλλογής δεδομένων. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις οι οποίες τους απευθύνθηκαν. It's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 I'm sorry Λοιπόν, ανάμεσα σε άλλα έθεσα και το θέμα καλύτερων κλοβών για τις οτόκες όρνηθες. Στις δύο τελευταίες ε, συναντήσεις του, των Υπουργών Γεωργίας και ζήτησα από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν τις πληροφορίες οι οποίες ε, ελείπουν. Κάποια κράτη-μέλη ανταποκρίθηκαν στην εκκλησία μας αυτή, κάποιες άλλες χώρες όμως ε, δεν έχουν ακόμα απαντήσει. Οι γεωργοί οι οποίοι έχουν επενδύσει στην ευημερία των ζώων του δεν θα πρέπει να τεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω της αδράνειας των υπολείπων γεωργών. Και τέλος να πω ορισμένα για την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων με την οποία ασχολείται και η Επιτροπή σας. Εγώ παρακολούθησα τη διαδικασία υιοθέτηση ε, της ε, έκθεσης Lines. Ε, τέθηκε και το θέμα της αναλογικότητας των εθνικών μέτρων και της σωστής πληροφόρησης ε, των παραγωγών σχετικά με την προσαρμογή των περιορισμών καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Αυτό σχετίζεται με την προσπάθεια η πρόταση αυτή να καλύψει όλες τις ανάγκες. Ε, παρατήρησα όμως ότι ορισμένες τροπολογίες σχετίζονται με συγκεκριμένα άρθρα της ε, τροπολογίας 2018 και της 26Β σχετικά με τις δυνατότητες των κρατών μελών να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τις καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων. Εμείς θα θέλαμε να υπάρξουν πιο στοχευμένες τροπολογίες για την κάλυψη ορισμένων κρατών που επιθυμούν τις ρήτρες opt-out εξαίρεσης. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή Περιβάλλοντος ψήφισε τις ε, τροπολογίες της έκθεσης Δελπάζ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά συνέπεια θα συνεχίσει τη συζήτηση των τροπολογιών που υιοθετήθηκαν πάντα έχοντας σαν στόχο την στενή συνεργασία με τους συνομοθέτες μέχρι το τέλος της διαδικασίας υιοθέτησης της πρότασης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Περιμένω τώρα πλέον και τις απόψεις σας και να μπορέσω να δώσω και τις απαντήσεις που ίσως θέλετε όπως μπορείτε. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο, σας ευχαριστούμε για την ε, πληρέστατη παρουσίαση. Το πρόγραμμά σας είναι πολύ πλούσιο και έχει πολύ σημαντικές ε, συναντήσεις και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για την Επιτροπή μας, ε, την Επιτροπή Γεωργίας. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε από τους συντονιστές, επομένως θα δώσω το λόγο απευθείας στον Άλμπερτ για να παρέμβει πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Επίτροπο. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας και από την προηγούμενη θητεία θα πρέπει να πω ότι είσαστε από τους Επίτροπους εκείνους που ε, εξαιρετικά συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ προσωπικό Έχω πολύ καλές εμπειρίες και από εσάς και από την Επιτροπή σας. Προκειμένου να μην υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των κρατών μελών. Ξέρετε φυσικά τι εννοώ για τα θέματα που αναφέρατε. Είσαστε υπεύθυνο αρμόδιο για ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα υγεία και πολιτική για του καταναλωτέ ε, μα ε, επηρεάζουν ιδιαίτερα στην Επιτροπή μα. Θεωρώ ότι κινούμαστε προ σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τι προδιαγραφέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την περαιτέρω εναρμόνιση του προκειμένου να μην υπάρχουν στρεβλώσει του ανταγωνισμού. Θίξατε επίσης και το θέμα των ελέγχων. Εδώ να υποδείξω ότι αυτό μπορεί να ξεπερνάει και τον τομέα αυτό, αλλά είναι σημαντικό να μιλήσουμε με την Επιτροπή, με τον Επίτροπο Εμπορίου, γιατί προγραμματίζονται συμφωνίες εμπορικές και με τις χώρες Μερκοσούρ. Στην προηγούμενη θητεία εφαρμόσαμε ε, πολύ αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία των φυτών εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να επιμείνουμε να εισάγονται μόνο προϊόντα τα οποία θα πληρούν τα δικά μας πρότυπα ασφάλειας. Γιατί δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στους γεωργούς πώς απαγορεύονται κάποια στοιχεία, κάποιες ουσίες για την προστασία των φυτών, αλλά παράλληλα εισάγονται προϊόντα από περιοχές όπου εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτές τις ε, ουσίες. Το ξέρω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με συμφωνίες του ΠΟΕ, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να καταλήξουν και να τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο οι συμφωνίες του ΠΟΕ προκειμένου να πληρούνται οι τα δικά μας πρότυπα. Πολλές φορές το έχω αναφέρει και έχω παραθέσει και αυτό που είχε πει ο Χέλμαν Κόλ ότι θέλουμε για ε, την προστασία των φυτών για τις ουσίες αυτές να ισχύουν τα ίδια που ισχύουν για τις εισαγωγές αυτοκινήτων. Αν θέλουμε να εισάγουμε ασιατικά αυτοκίνητα, να πληρούν τις δικές μας προδιαγραφές ασφάλειας. Έμα το ίδιο θέλω και για την εισαγωγή τροφίμων και την εισαγωγή ζωοτροφών. Να εισάγονται μόνο εφόσον ανταποκρίνονται στις δικά μας πρότυπα ασφάλειας σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων, ο ίδιος ο Γεωργός, ο έχει συμφέρον να εφαρμόσει τις σχετικές προδιαγραφές που αποβαίνουν προς όφελος των ζώων. Αναφέρετε διάφορα στοιχεία, να σας, σας παρακαλέσω να είναι εφαρμόσιμες αυτές οι διατάξεις. Γιατί παλιά δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε τα θέματα ε, για την μεταφορά των ζώων. Δηλαδή, ενώ επί δεκαετίες ε, μπορούσαμε να μεταφέρουμε εκτροφή στα ζώα 50-60 χιλιόμετρα, πλέον είχαν αλλάξει οι κανόνες και αυτό ήταν πραγματικά ακατανόητο για τους εκτροφεί. Και τέλος, μιλήσατε και για απλούστευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα μέτρα τα οποία προγραμματίζετε και τα οποία επιθυμείτε να εφαρμοστούν να παραμείνουν όσο το δυνατόν απλούστερα, να μην ε, επιβάλλουν καινούργια γραφειοκρατία, αλλά από πλευράς διοικητικής να είναι εύκολα εφαρμόσιμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το μελλοντικό σας έργο. Ευχαριστώ. Ο Λουίς Καπούλα Σάντορς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την παρουσίασή σας και συμφωνώ απολύτως με τις προτάσεις ε, που μας παρουσιάσετε για το πρόγραμμα εργασίας και μάλιστα ελπίζω να μπορέσετε και να τις ε, υλοποιήσετε επιτυχώς. Δύο ερωτήσεις. Τη μία την έθεσε ήδη ο συνάδελφος Ντες και είναι το θέμα του ελέγχου στα σύνορα. Ο Επίτροπος είπε ότι θα μπορούσαν να γίνουν βελτιώσεις στο σύστημα εάν τα υγειονομικά όρια είναι τα τελευταία μας όρια και θα πρέπει να υπάρχει και αμοιβαιότητα στις απαιτήσει προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό για τους ε, γεωργούς και κτηνοτρόφους μας. Όπως είπε ο κύριος Ντέσκ, ε, το υποστηρίζω και εγώ, μακάρι να μπορέσετε να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα πώς μπορείτε να βελτιώσετε τους ελέγχους. Δεύτερη ερώτηση κύριε Πρόεδρε, στην παρουσίασή σας δεν θίξατε το ζήτημα, αλλά είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας και πρόκειται για τη χρήση ηχθιαλεύρων και τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε και τι εξέλιξη βρέπετε για τη χρήση αυτών των ε, προϊόντων, ε, διότι υπάρχει πίεση και από την κοινή γνώμη και από τους ε, διάφορους τομείς που χάνουν ανταγωνιστικότητα με τη χρήση αυτών των κανόνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και μας εξηγήσατε το πρόγραμμά σας για το τρέχον έτος. Τρία στοιχεία θα ήθελα να τονίσω. Αναφέρατε σε ό,τι αφορά την υγεία των ζώων, την ταυτοποίηση. Όπως τα ξέρετε, η εφαρμογή για την ταυτοποίηση των ε, αμνών έχει προκαλέσει μεγάλη δυσκολία και μεγάλη διαμάχη από πρακτικής άποψης ε, σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους να σας ρωτήσω. Λοιπόν, θα γίνει μία αναθεώρηση σε κάποια φάση του κανονισμού για να ε, καθορίσουμε κατά πόσον ε, υπάρχουν όντως τα πρακτικά αυτά προβλήματα και πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι διαδικασίες με καλύτερο τρόπο. Σε ό,τι αφορά και τα μεγάλα κοπάδια στη Σκωτία, Φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι από την Ιρλανδία έχουν ε, προβλήματα. Το θέμα λοιπόν παραμένει η πρακτική εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Μιλήσατε επίσης για ένα νόμο για την ευημερία των ζώων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και πάλι θα ήθελα να δεσμευτείτε σε ό,τι αφορά τα πρώτα σας σχόλια είπατε ότι θέλετε να υπάρξει μια εναρμόνιση σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για τη μεταφορά των ζώων. Ε, θα ήθελα να μου εγγυηθείτε ότι εκεί θα επικεντρωθείτε, γιατί υπάρχει γενικά η αντίληψη στη χώρα μου του κλάδου ότι δεν χρειαζόμαστε πιο πολλούς νόμους, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι η καλύτερη εφαρμογή των ειδηφιστάμενων νομοθεσιών. Θα ήθελα λοιπόν να μου εγγυηθείτε ότι αυτό θα ακολουθήσετε ως κατευθυντήρια γραμμή. Τέλος, μιλήσατε για, τους, τα κλουβιά. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένο το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Είπατε ότι θέλετε να διασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη ακολουθούν συμβατές πρακτικές. Οχτώ μήνες όμως παραμένουν μέχρι την ημερομηνία και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, έχουμε 80 εκατομμύρια αυγά που δεν είναι συμμορφωμένα με τη διαδικασία αυτή. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Προφανώς δεν αρκεί ο προγραμματισμός για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε μέχρι 1η Ιανουαρίου του 2012. Τι σκοπεύει να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις και τι θα κάνετε. 80 εκατομμύρια αυγά δηλαδή θα είναι ξαφνικά παράνομα από πρώτες πρώτες του 2012. Εκατομμύρια λίρες έχουμε εξοδέψει για να συμμορφωθούμε με το σύστημα και θα συνεχίσουμε να έχουμε μειονέκτημα συγκριτικά με άλλους που δεν έχουν εφαρμόσει τα συστήματα αυτά. Ο κύριος Χόουσλινγκ. Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που ήρθατε εδώ. Ε, να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, για θέματα τα οποία δεν αναφέρατε. Ένα θέμα το ανέφεραν και οι συναδελφοί. Είπατε, ε, αναφέρατε τα περί πρωτεϊνών ε, ζωικών τι ακριβώς σχεδιάζεται, γιατί εμείς έχουμε τοποθετηθεί με σαφήνεια ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες. Εσείς τι προβλέπετε. Ύστερα, δεν έχει περάσει πολύ καιρό στη Γερμανία από το σκάνδαλο με τις διοξίνες. Τι έχετε πετύχει σε, ως προς το θέμα αυτό στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Τι γίνεται με την ε, κυβέρνηση στη Γερμανία και γιατί είστε τόσο κατηγορηματικός κατά μία θετικής λίστας, ενό θετικού καταλόγου. Έλαβα τη σχετική σας επιστολή. Τρίτη ερώτηση για την κλωνοποίηση. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, εσείς πλέον ε, έχετε τη σκητάλη για να υποβάλλετε μια νέα πρόταση. Θα υποβάλλετε γρήγορα κάποια πρόταση ή σε πρώτη φάση θα προτιμήσετε να ακολουθήσετε άλλες οδούς. Γιατί νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων να συζητήσουμε το θέμα αυτό και στο κοινό ψήφισμα. Συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ε, επικίνδυνων φυτών και των γενετικά τραποποιημένων φυτών. Αλλά ρωτώ, είχατε πει πέρσι ότι εξακολουθείτε να είσαστε υπέρ ε, μηδενικής ανοχής σε ό,τι αφορά τους σπόρους. Ελπίζω να μην αλλάξετε γνώμη και ελπίζω να μην κινδυνεύουν οι σπόροι. Να εξακολουθείτε να υποστηρίζετε τη μηδενική ανοχή. Και τι γίνεται με την εισαγωγή ζωοτροφών. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα τι ποσοστό των ζωοτροφών επιστρέφεται τα τελευταία χρόνια επειδή διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκμόλυνση. Δεν έχουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, ποτέ πάντα ακούμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό για τις, ε, για τις εωτόκους όρνηθες. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε το θέμα. Αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και είναι όλο και πιο κατεπήγον το ζήτημα. Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει σωστή εφαρμογή. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πιεστικά τα ερωτήματα και περιμένουν οι κτηνοτρόφοι από εμάς κάποια απάντηση για τα γεννητικώς τροποποιημένα φυτά τώρα και πάλι. Να επανέλθω στο θέμα αυτό. Μας εξηγήσατε την καινούργια νομοθεσία, αλλά εξακολουθούν να ανακύπτουν πολλά ερωτήματα. Στην Ευρώπη, πώς έχουμε προχωρήσει για μια κοινή ε, ευθύνη, τι γίνεται με τη μεταρρύθμιση της ΕΦΣΑ, και πότε θα υπάρξουν ε, παρόμοιοι κανόνες, ίδιοι κανόνες ε, για την ε, σπορά. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και νομίζω ότι θα πρέπει να μην τα αφήσουμε μόνο στα χέρια των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον. James. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα περισσότερα από τα θέματα που ήθελα να θέξω έχουν ήδη αναφερθεί από τους προλαλήσαντες επομένως θα είμαι λακωνικός. Για τους κλοβούς ε, των ορνηθών, ε, λέτε ότι ε, κάποια κράτη-μέλη δεν απαντούν και προσπαθείτε να δείτε αν μας απαντούν. Αυτοί όμως που έχουν συμμορφωθεί μήπως βρίσκονται σε μειονεκτική θέση πλέον. Και θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε, διότι εκπνέουν και οι προθεσμίες. Αρχίζουμε να φτάνουμε κοντά στα περιθώρια και θα ήθελα να γνωρίζω τι θα γίνει, διότι θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας επί του θέματος, καθώς συμφωνώ και με αυτό που μας είπατε. Αυτοί που έχουν ε, επιτύχει και έχουν ανταποκριθεί σε αυτό που τους ζητήθηκε, δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτή τη στιγμή, είναι αδύνατον. Διότι δεν μπορούμε να επιδονώσουμε εμείς τη θέση τους. Για τη Μερκοσούρ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Άλμπερτ. Συνήθω οι επίτροποι όταν αναφέρονται, αναφέρονται σε παρόμοιε προδιαγραφές και όχι στις ίδιε προδιαγραφές πλέον. Και νομίζω κύριε επίτροπε ότι παρόμοιες και ίδιε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό που σας λέω λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να είναι ε, πανομοιότυπες οι προδιαγραφές. Δεν μπορείτε να περιμένετε οι παραγωγοί στην Ευρώπη να πληρούν τις προδιαγραφές που τους απαιτούμε, να δίνουμε τα στοιχεία αυτά στον καταναλωτή και μετά να εισαγάγουμε στοιχεία κατωτέρων προδιαγραφών. Παρόμοιες προδιαγραφές δεν είναι αποδεκτές. Θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες επακριβώς προδιαγραφές. Εχθές στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, συζητήθηκε ε, το θέμα των ζωικών αλεύρων και εγώ είμαι και σκιώδης εισηγητής. Ένας συνάδελφος ε, είπε ότι οι απαντήσεις μου στο θέμα αυτό είναι συναισθηματικές. Εγώ όμως είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου ζήσαμε όλη την τραγωδία για τη σπογκώδια εγκεφαλοπάθεια. Και γνωρίζω και τα επιχειρήματα για τα ζωικά αλευρά, θεωρείται ότι είναι πρωτεΐνη που βοηθά ε, για την εκτροφή των χείρων και άλλων ε, ζώων γιατί δεν έχουμε επαρκή σόγια και ίσως είναι και μια κατάλληλη λύση. Αλλά πρέπει να σας πω και νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο Λίς Πούλα Σάντον σε αυτό, οι καταναλωτές θα θέλουν να γνωρίζουν όταν χρησιμοποιηθούν ζωικά αλευρά κατά πόσο είναι απολύτως ασφαλή και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν λέμε απλώς ότι επιστημονικός είναι ορθό, θα πρέπει να υπάρχει μια παρουσίαση της άποψη αυτής και θα πρέπει να συμφωνήσει μαζί σας και το κοινό, διότι θεωρώ ότι θα υπάρξει μεγάλος βαθμός ε, ε, και... Ε, έλλειψης εμπιστοσύνης και διαφωνίας επί του θέματος. Και ξέρετε κιόλας ότι ο κίτρινος τύπος θα παρουσιάσει ένα σωρό δημοθεύματα και θα το μεγαλοποιήσει το πράγμα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ε, με μεγάλη ευαισθησία. Δεν θεωρώ ότι είναι κακή ιδέα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ, James. Προχωράμε τώρα. Μίλησαν όλοι οι συντονιστές. Α, όχι, ο Λορέντζο δεν μίλησε. Μετά το Λορέντζο, λοιπόν, θα περάσουμε στου υπολείπου και θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο σύντομοι, γιατί είναι μεγάλος ο κατάλογος. Θα είμαι σύντομο, συνάδελφοι, γιατί τα είπαν και οι συνάδελφοι αυτά που ήθελα να πω. Θεωρώ, ακούγοντας και τους συναδέλφους συντονιστέ, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους. Θέλουμε τα εμπορεύματα τα οποία εισάγονται στην Ευρώπη να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητες με τα δικά μας προϊόντα και για τους καταναλωτές αλλά και για να μην υπάρχει αθέμιδος ανταγωνισμός ε, στις ξένες εισαγωγές. Περιμένω λοιπόν και μια απάντηση για συγκεκριμένες λύσεις επί του θέματος. Κατανοώ ότι δεν είναι εύκολο το ζήτημα, πρόκειται για μια μάχη ε, η οποία είναι πολύ επίκαιρη, αλλά θα πρέπει να βρούμε κοινό τόπο μεταξύ των διαφόρων επιτροπών, ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό που συμβαίνει επανειλημμένως και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ Λορίνζο. Ο κύριος Χάσφορντ έχει το λόγο και μετά κυρία Πόλσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τα σχόλια που έκανε. Δύο συγκεκριμένα στοιχεία θα ήθελα να θίξω. Πρώτο, σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, όπου θα ξέρετε φυσικά ποιε είναι οι προτάσεις οι σχετικές. Χρησιμοποίησατε την, τον όρο αναλογικότητα Συγκεκριμένα, αυτό που θα ήθελα να θίξω είναι το εξή. Η δυσκολία που θα αντιμετωπίσετε για να εξισορροπήσετε τα εμπορικά συμφέροντα των ε, ε, εταιριών εκτροφής και των προδιαγραφών για την ασφάλεια των φυτών. Και ιδιαίτερα για να μειώσετε το κόστο για τους αγρότες. Ρωτώ λοιπόν, ποια είναι η στάση σας και ποιες είναι οι προτάσεις σας οι νομοθετικές και ρυθμιστικές σε ό,τι αφορά τους ε, σχετικούς ε, σπόρους που έχουν αποθηκευτεί. Ξέρω ότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα γενικά. Ιδιαίτερα όμως σε ό,τι αφορά τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς θα αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβλημα και υποπτεύομαι ότι θα πρέπει να το έχει αυτό στην ατζέντα της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άλλο ζήτημα τώρα το οποίο σας έχω γράψει κιόλα έχει να κάνει με, την, ε, με τις εξωτερικές ε, περιοχές και την... Ε, να σας πω ότι έχουμε μία περιφέρεια, μία περιοχή στην περιφέρειά μας όπου αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερε δυσκολίες και δεν μπορούμε να, να ανταποκριθούμε στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά το αγροτικό απόθεμα. Έχουμε γράψει και σχετική επιστολή. Αυξάνεται λοιπόν το κόστος ακριβώς στις πιο δύσκολες ε, περιοχές αυτές και τελικά καθιστά μη φιώσιμη η διατήρηση αυτού του αποθέματος. Οι τοπικές αρχές δεν προτίθενται να χρηματοδοτήσουν και ψάχνουμε κάποιο τρόπο να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Η κυρία Πόλσον, η Αντιπρόεδρος και μετά ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Η παρουσία σας εδώ δείχνει ότι ενδιαφέρεστε για τα θέματα τα οποία συζητάμε. Δεν θα επανέλθω σε όλα τα θέματα τα οποία αναφέρατε και στις ερωτήσεις που ήδη τέθηκαν. Το θέμα είναι αν μπορούμε να βρούμε ένα επίπεδο προστασίας της ε, ε, υγείας των ζώων επαρκές. Απαιτείται να υπάρξει ένα κοινό σύστημα ελέγχου. Αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ποιος είναι ο κανόνας που ισχύει στην Ευρώπη σήμερα, γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις εθνικές ρυθμίσεις όχι μόνο τις νομοθετικές εθνικές ρυθμίσεις, αλλά και τις πρακτικές και τις μεθόδους που ακολουθούνται. Συνεπώς, θα πρέπει η νομική ρύθμιση από τη μία, το κείμενο του νόμου δηλαδή και η πρακτική από την άλλη να ενιοποιηθούν. Τώρα το σύστημα που βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα στο σύνολο της τροφιμικής αλυσίδας. Αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί. Όταν το επίπεδο έκθεση σε κίνδυνο, όταν το επίπεδο κινδύνου αν θέλετε, δεν είναι σαφές ποιο είναι και δεν είναι κατανοητό για τους ίδιους τους τοπικούς επιθεωρητές, τους τοπικούς ελεγκτές που καθημερινά θα πρέπει στην πρακτική, στη ρουτίνα να κάνουν τους ελέγχους, τότε τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα γιατί και εδώ έρχεται και το θέμα των διαφορετικών μεθόδων που ακολουθούνται. Εδώ δημιουργούνται περαιτέρω κίνδυνοι και δημιουργείται ουσιαστικά μια θα έλεγα στρεβλή μορφή ανταγωνισμού στο εσωτερικό της, της αγοράς μας. Είναι απαραίτητο και οι κανόνες από τη μία αλλά και οι πρακτικές από την άλλη να είναι συγκρίσιμες. Εφόσον το πετύχουμε αυτό, τότε μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά και για τα θέματα των εισαγωμένων προϊόντων. Πρέπει να δούμε ποια είναι η εσωτερική αγορά και να βεβαιωθούμε ότι οι διαφορές στο εσωτερικό της εσωτερικής αγοράς δεν είναι τεράστιες ε, ε, για τομείς ε, που καλύπτονται από νομικές ρυθμίσεις. Πρέπει να είμαστε πιο σαφείς και πιο αυστηροί όταν προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ανάλυσης των κινδύνων. Ένα άλλο θέμα είναι ο τρόπος ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να να αξιολογήσουμε τη μέθοδο που ακολουθήσαμε για το εμβόλιο Blue Tongue. Σχετικά με το συγκεκριμένο εμβόλιο και σχετικά με τον αυθόδη γενικότερα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να προλαμβάνουμε και όχι να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες εκ των υστέρων. Ταραμπέλα. Καλημέρα σας Επίτροπε. Από την 3η 29 το πρωί γνωρίζουμε ότι είστε πλέον υπέρ της κλωνοποίησης των ζώων και του κλωνοποιημένου κρέατος. Μιλάτε σωστά για την υγεία βέβαια των ανθρώπων και των ζώων και θα ήθελα η συμπεριφορά σας να ανταποκρίνεται στα λεγόμενά σας. Γιατί λοιπόν στις 29 Μαρτίου το πρωί κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο για τα κλωνοποιημένα κρέατα, από ό,τι μου είπαν, και δεν ήμουν εγώ εκεί, αλλά η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ με την κυρία Τεστόρη, η οποία ήταν ιδιαίτερα έμονη, και με τον υπερφιλελεύθερο Επίτροπο Ντεγκούχτ, είπαν ότι ήταν υπέρ της εμπορίας του κλωνοποιημένου κρέατος παρά τις επιθυμίες του Ευρωπαίου καταναλωτή, παρά τι επιθυμίε ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαγορεύοντας μάλιστα και την ετικετοθεσία που θα ενημέρωνε τον καταναλωτή για το τι καταναλώνει. Από τη μία λοιπόν καλείστε να υπερασπιστείτε τους Ευρωπαίους καταναλωτές και από την άλλη να προωθήσετε τις απόλυτα εμπορικές πρακτικές οι υπερφιλελεύθεροι του εμπορίου θριαμβεύουν μέχρι τώρα. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Επίτροπε να μου πείτε αν στο μέλλον θα υπερασπιστείτε πράγματι τον καταναλωτή σε σχέση με τις επιθυμίες του καταναλωτή και σε σχέση και με τις αντιφάσεις οι οποίες μας χαρακτηρίζουν, αναφέρθηκε η κυρία Πόλσεν σε αυτό, και τις υπερφιλελεύθερες μερικές φορές σχιζοφρενικές αντιλήψεις ορισμένων συναδέλφων. Βλέπουμε ότι επιβάλλονται σκληροί κανόνες στους παραγωγούς μας, αλλά ανοίγουμε το εμπόριο και την εμπορία προϊόντων σε οτιδήποτε πλέον. Και μας οδηγείται στο να αποδεχθούμε πράγματα απαράδεκτα, τα οποία ο Ευρωπαίος καταναλωτής έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί. Λεφόλ και μετά Μποδέ. Δύο σύντομα λόγια. Καταρχάς να συμφωνήσω ε, περίπου με τον Μάρκ Ταραμπελά. Πρέπει να είμαστε ε, πολύ επιφυλακτικοί για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη τοποθετείται στη διεθνή σκηνή και εσωτερικά όταν πρέπει να πάρει αποφάσεις σχετικές με την προστασία του καταναλωτή. Δεν μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές πρακτικές και διαφορετικές πορείες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίπεδο διμερών σχέσεων θέτει ρήτρε κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Είστε υπέρ των ρητρών αυτών, θα υπερασπιστείτε τις θέσεις αυτές ή δεν θα το κάνετε αυτό. Το δεύτερο αφορά τα γενετικά τροποποιημένα. Έχει γίνει προσπάθεια και στη δική μας Επιτροπή, η οποία λήφθηκε υπόψη και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της τροπολογίες της και θα ήθελα να μάθω ποια είναι η κατάσταση σε επίπεδο Συμβουλίου και σε επίπεδο Επιτροπής. Θα υποστηρίξετε την θέση η οποία ελπίζω να ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση των κανόνων και των συνθήκων στα πλαίσια των οποίων τα κράτη δεν θα χρησιμοποιούν ή μπορούν να αποφασίσουν να μην χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένη σπορά. Ευχαριστώ Επίτροπε. Τρία σημεία, μία παρατήρηση σε σχέση με αυτά που είπε ο Μάρκ Ταραμπελά. Είπε πράγματα σωστά. Αλλά θα ήθελα να προειδοποιήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην ξαναζήσουμε αυτά που είδαμε το 1980 όταν είχε θελήσει να επιβάλλει τις ορμόνες στην ακτινοτροφία και είχε οδηγηθεί τότε σε μποϊκοτάζ η αγορά των προϊόντων των καταναλωτών. Όταν υπάρχει κίνδυνο στην αγορά τότε φοβάμαι ότι θα προκληθούν τεράστιες αντιδράσεις και τα πρώτα θύματα θα είναι οι ίδιοι οι οι οποίοι θα δουν την αγορά τους να περιορίζεται και να καταστρέφεται. Γι' αυτό λοιπόν προς το συμφέρον των γεωργών σας ζητώ να είστε κατά της εισαγωγής κλωνοποιημένου κρέατος. Τρεις παρατηρήσεις τώρα. Η πρώτη αφορά την νομοθετική ρύθμιση την οποία προτείνεται. Άκουσα τις προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος με την ψηφοφορία της σήμερα το πρωί και θα ήθελα να σας πω επίσημα σε εισαγωγικά σήμερα ότι εγώ θα είμαι υπέρ των προτάσεων αυτών. Εγώ ήμουνα κατά της εθνικοποίησης των γενετικά τροποποιημένων, αλλά θα συμφωνήσω με την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος εφόσον μπορέσουμε να δείξουμε ότι πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο. Το σύνολο των στοιχείων τα οποία εμείς μας δώσατε σχετικά με την αποδοχή, απόρριψη των γενετικά τροποποιημένων είναι σωστά στοιχεία, είναι ζωστοί κανόνες εφόσον περάσουν μέσα από το φίλτρο της αναθεώρησης του 2012. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία μπορεί να χρησιμεύσουν στη συνολική ανάλυση της κατάστασης των γενετικά τροποποιημένων και θα σας στηρίξω και επίσημα στην προσπάθεια την οποία κάνετε και θα κάνετε από εδώ και πέρα. Δεύτερον, για τη σπορία. το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Εδώ θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχει μηδενική ανοχή στα γενετικά τροποποιημένα στη σπορία. Δεν είναι φιλοσοφικό το θέμα, δεν είναι δεοντολογικό το θέμα. Είναι απλά θέμα πολλαπλασιαστή. Εάν δεχθούμε έστω και 0,1% σε μία φάση, τον επόμενο χρόνο είμαστε στο 0,5% και μετά είμαστε στο 1% και μετά είμαστε στο 3% και πάει λέγοντας. Οπότε θα υπάρξει μία σταδιακή επιμόλυνση του συνόλου των διαθεσίμων σπόρων. Τρίτο στοιχείο και θα σταματήσω εδώ αφορά τους λεγόμενους γεωργικούς σπόρους, τους σπόρους των γεωργών. Ξέρετε ότι το 2010 η οργάνωση του Παγκόσμια των Τροφίμων αναγνώρισε τη σημασία της βιοπικιλότητας της σποράς στην γεωργική παραγωγή. Τίθενται θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη μία και τίθενται και θέματα ελευθερίας χρήσης από την άλλη. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ένα ανάμεικτο σύστημα το οποίο ενισχύει τις μεγάλες επιχειρήσεις εις βάρος των δικαιωμάτων των γεωργών να χρησιμοποιούν εκ νέου την δική του σπορά. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Η Ευρώπη επέλεξε το δικό της σύστημα και ήταν καλό που επέλεξε το δικό της σύστημα, αλλά δυστυχώς σήμερα πολλές επιχειρήσεις προσθέτουν νέες ευρεσιτεχνίες με γενετικά τροποποιημένα κτλ. Συνεπώς ε, και στα πλαίσια της ΕΦΣΑ θα γίνουν συζητήσεις για τις νέες βιοτεχνολογίες. Θα πρέπει να καταλήξουμε κάπου για το πώς θα προστατεύσουμε τη γεωργική σπορά η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ιδιαίτερα σε νέες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Πολωνία. Ευχαριστώ. Κυρία σε ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι που ήρθατε εδώ σήμερα για να συζητήσετε το πρόγραμμα εργασίας σας. Ένα, ε, μια ερώτηση να κάνω. Μιλήσατε για συλλογή δεδομένων. Τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα συλλέξει τα δεδομένα αυτά. Θα αποφύγουμε μια διπλή συλλογή δεδομένων, προκειμένου να είμαστε αποδοτικοί και αποτελεσματικοί. Γιατί τα δεδομένα αυτά δεν αρκεί να τα μαζέψουμε, θα πρέπει να αξιολογηθούν και σωστά και αυτό θα προκαλέσει φόρτο εργασία. Επίσης να πω ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις κυρίως είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές ως επιτοπλίστων. Και αν μετά την εργασία τους για την γεωργία, τα κερδικά του καθήκοντα πρέπει να κάτσουν να μαζέψουν και να συλλέξουν και στοιχεία, θεωρώ ότι αυτό θα τους ε, επιβάλλει υπερβολικά, μεγάλο φορτό. Και τι γίνεται θα, με τα στοιχεία αυτά, με τα δεδομένα αυτά. Θα συγκεντρωθούν σε μια τράπεζα δεδομένων. Πώς θα προστατευτούν προκειμένου να μην έχει ο καθένας πρόσβαση σε αυτά. Προκειμένου να μην έχουν ε, αγωνιστικό μειονέκτημα Γεωργή, με τη συλλογή των δεδομένων αυτών. Γιατί αν ε, τα ανοίξουμε σε όλους τα στοιχεία αυτά, θα μπορούν να τα κοιτάξουν και άλλες επιχειρήσεις και θα μπορούσαν ε, ενδεχομένως να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Επίσης, δείξαμε το θέμα των οτόκων ορνηθών. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Έχει το θάρρος και την τόλμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την απαγόρευση της χρήσης των κλοβών να κλείσει τις επιχειρήσεις που δεν θα συμμοφορθούν. προκειμένου όντω να υπάρξει πλεονέκτημα για όσους έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις. Κάτι άλλο τώρα για τη μεταφορά των ζώων. Θα ληφθεί υπόψη άμα η μελλοντική συγκέντρωση σφαγίων και ενδεχόμενη έλλειψη σφαγίων. Τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι δυνατόν αφενός να περιορίζουμε χιλιομετρικά τη μεταφορά και αφετέρου να μην υπάρχουν σφαγεία σε ολόκληρες περιοχές. Τι θα κάνουν οι γεωργοί, οι εκτροφοί, συγγνώμη. Äh, Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω κύριο Γιάρ, να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο που ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας. Μία ερώτηση να κάνω, γιατί πολλές ερωτήσεις έκαναν ήδη οι συνάδελφοι. Να ρωτήσω. Είχαμε και μια αλληλογραφία αναφορικά με το θέμα αυτό και μου είπατε ότι βρίσκεται στη φάση συζήτηση για τις μετακρατημέλη, για τις ε, και μας είπατε ότι κάποια κράτη-μέλη δεν συνεργάζονται απαραίτητα και φαντάζομαι ότι αυτά είναι τα κράτη τα οποία έχουν προβλήματα με την εφαρμογή. Αυτά τα κράτη θα δείξουν ε, λιγότερο πνεύμα συνεργασίας. Να συμφωνήσω λοιπόν με την κυρία Ράιμερς. Ποιο είναι το ε, εναλλακτικό σας σχέδιο, τι θα γίνει με τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν είναι σε θέση εμπρόθεσμα να εφαρμόσουν το σχετικό κανονισμό για τις οτόκους ορνηθές. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία για το θέμα αυτό. σε ό,τι αφορά την απαγόρευση αυτή. Έχουμε ξεκινήσει από πολύ πιο πριν και έχουμε χάσει μεγάλο τμήμα της αγοράς εξαιτίας της αλλαγής αυτής.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 Um, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, οδηγία για τις οτόκες όρνηθες. Ίσως θα έπρεπε να δούμε και πόσα κράτη-μέλη έχουν αποστείλει τις πληροφορίες και επομένω και ποιοι δεν αποστέλουν πληροφορίες για να ξέρουμε κατά πόσο χρειαζόμαστε ένα εφεδρικό σχέδιο καθώς οι συνάδελφοι θεωρούν ότι χρειαζόμαστε. Ε, συμφωνώ με τα σχόλια για την νομοθεσία για τη μεταφορά των ζώων και ζητώ να εφαρμόσουμε την νομοθεσία που έχουμε και να μην προσπαθήσουμε να ε, νομοθετήσουμε εκ νέου, διότι γελιοποιούμεθα στα μάτια των καταναλωτών και των κτηνοτρόφων και παγκοσμίω άλλωστε, αν ακολουθούμε τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Όσον αφορά του ελέγχου των εισαγωγών, μας δώσετε διεξοδικές πληροφορίες επί του θέματος. Να ρωτήσω το εξή απλό. Ε, θεωρείτε την παρούσα κατάσταση για τους ελέγχους, ε, για τις εισαγωγές. Είναι ικανοποιητική, μη ικανοποιητική. Διότι θα έπρεπε να γνωρίζουμε γιατί και εμείς ανησυχούμε και τις εξέφρα, ε, σε τις ανησυχίες μας ο κύριος Ντές για τους ελέγχους στα σύνορα. Επίσης, θα μπορούσατε να μας συνοψίσετε τις επιπτώσεις της, ε, του γεγονότος ότι δεν μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε για ένα νέο κανονισμό για τα νέα τρόφιμα, για τα novel foods εγώ δεν ξέρω σαφώς τι επιπτώσεις έχει αυτή η αποτυχία και τι ακριβώς με λιγενέστε. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα προσωρινό πρόεδρο, έχουμε κενό στην Προεδρία τα τελευταία πέντε λεπτά, αλλά η δημοκρατία λειτουργεί αποτελεσματικά. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να μας θεωρήσετε ως συμμάχους σας εδώ στην Επιτροπή μας ε, και εδώ διακυβεύεται και η δική σας αξιοπιστία και η δική μας. Έχω συζητήσει με ε, υπαλλήλου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να το προχωρήσει στα άκρα, αλλά και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε και θέλουμε να εφαρμόζονται και να τηρούνται οι νόμοι που έχουμε ψηφίσει. Έχω κάποιες παρατηρήσεις ε, για τις ευρωπαϊκές ταυτότητες των ζωηδών θεωρούμε ότι είναι μια χρήσιμη τεχνολογία και είναι ένας τρόπος διαχείρισης των αποθεμάτων ε, και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με την εφαρμογή θα ήθελα να γνωρίζω και κάποια πράγματα ε, για τον οδικό χάρτη για το TSE η επιστήμη έχει προχωρήσει και ίσως είναι και η ώρα να ε, κάνουμε και εμείς πιο αυστηρούς κανόνες για την τήρησή του. Υπάρχει το θέμα του αυστηρού κλίματος, της συγκεκριμένης γεωγραφίας και ε, νομίζω ότι είναι αποτελεσματικά αυτά και για κάποια νησιά στη Σκωτία και νομίζω ότι εδώ ε, υπάρχει λόγος να τηρήσουμε και εμείς τους κανόνες. Και κάτι πιο τεχνικό, θα γνωρίζετε από την αλληλογραφία που είχαμε αρκετοί από εσά ότι υπάρχουν συζητήσεις της ΚΟΦΚΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα πολλές από τις περιφέρειές μας, κυρίως τα Βρετανικά ε, νησιά. Οι Ιρλανδοί, οι Σκοτοί έχουν σοβαρά θέματα για τα θέματα της αδειοδότησης του προϊόντος. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι θα το εξετάσουν οι υπαλληλοί σα και δεν θα ε, παραμείνει κενό γράμμα. Υπάρχει εμπορική πραγματικότητα και θα πρέπει να ανταποκριθούμε και στις ανάγκες της ε, επιστήμης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και λυπάμαι που καθυστέρησα, αλλά δυστυχώ δεν εξαρτάται από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε εδώ, γιατί με προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση ω κτηνοτρόφο, ω ε, από ένα τμήμα της Ευρωβρετανία όπου υπήρξαν μεγάλες εξαγωγέ ότι μου λέτε ότι α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μα δεν με ακούτε όμως αυτή την ώρα και πολύ λυπάμαι, αλλά αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο δίλημα, γιατί φυσικά καταλαβαίνω τι λένε εδώ πέρα οι συνάδελφοι και ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Από 1η Ιανουαρίου θα πρέπει 100 εκατομμύρια ορνητές να βγουν από τα κλουβιά πώς θα εγγυηθούμε την ασφάλεια τους ή θα λέμε ότι 80 εκατομμύρια αυγά κάθε μέρα θα πρέπει να καταστρέφονται και να απορρίπτονται με ασφάλεια. Και αυτό προκαλεί και άλλο ένα πρόβλημα. Αυτά τα αυγά προορίζονταν για κάποια αγορά και οι Ευρωπαίοι θα εξακολουθούν να θέλουν να φάνε αυγά. Τι θα γίνει, θα, θα εξάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα τρώνε οι Ευρωπαίοι μάλλον θα εισάγονται τα αυγά αυτά και ποιος θα ξέρει τότε ε, τι προδιαγραφές θα πληρούν τα αυγά αυτά. Και επίσης ε, όλες αυτές οι όρνηθες που ε, θα αναγκαστούμε να ε, εκτελέσουμε από 1η Ιανουαρίου τελικά τι θα γίνει, τι θα έτρωγαν, θα έτρωγαν πλέον με τρόφιμα τα οποία ζωτροφές οι οποίες δεν θα χρησιμοποιούνται. Τι θα κάνετε λοιπόν για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Αγνιού, σας ευχαριστώ όλους. Και αυτή τη φορά αγαπητέ Επίτροπε, συλλέξατε πάρα πολλές ερωτήσεις και θα προσπαθήσετε τώρα να καλύψετε τις ευαισθησίες οι οποίες εκφράστηκαν από όλους τους συναδέλφους. Ο κύριος Ντάλι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Τα εξετίμησα δεόντως. Αυτές οι συζητήσεις ε, με βοηθούν εμένα προσωπικά και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι να κατανοήσουμε τις απόψεις, την αίσθηση που έχετε γενικά στο Κοινοβούλιο, τις προτεραιότητές σας και τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα οποία ακούστηκαν για το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης. Κατανοώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Εγώ θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η βασική μου ανησυχία είναι να προσπαθήσω να καταστήσω ε, ορθολογικές, απλούστερες και εναρμονισμένες τις ρυθμίσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω μας. <clears throat> Νομίζω ότι πριν από οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να αναλύσουμε το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την εφαρμογή αυτών των νομικών ρυθμίσεων που είναι σε ισχύ και να δούμε επίσης και ποιο είναι το περιθώριο το οποίο έχει κάθε, ε, κάθε ρύθμιση, ποιο είναι το περιφερειακό κόστος, ποιο είναι το περιφερειακό όφελος για το γεωργό, για την κοινότητα από την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων. Γενικά λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσουμε από τη διαδικασία αυτή. Από κοινού θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα απλουστεύσουμε και να καταστήσουμε τη γεωργία μας πιο ανταγωνιστική από τη σήμερα, χωρίς σε καμία περίπτωση να μειώσουμε εμείς τα επίπεδα ασφαλείας και τα επίπεδα ασφαλείας γενικότερα θα έλεγα για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Νομίζω ότι ο τομέας των τροφίμων είναι στην ουσία ο, βασικός φορέας της εσωτερικής αγοράς και της εικόνας της εσωτερικής αγοράς. Νομίζω ότι εμείς μπορούμε να παρέχουμε στον καταναλωτή καλά γνήσια προϊόντα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η προσβασιμότητα στα προϊόντα αυτά να είναι ε, θα έλεγα ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ένα από τα βασικά θέματα το οποίο τέθηκε είναι τα επίπεδα σε σχέση με τα επίπεδα εισαγωγών από τρίτες χώρες. Εγώ προσπαθώ να είμαι απλούστατο στον τρόπο που σκέφτομαι. Τα επίπεδα ασφαλείας τα οποία εμείς θέτουμε έχουν σαν στόχο να προστατεύσουν τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται από από όλα τα προϊόντα τα οποία πιθανώς εμφανίζονται στα ράφια των κατασκημάτων μας. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο όλα τα προϊόντα να είναι αυτά τα προϊόντα να είναι ασφαλή ανεξαρτήτως από πού προέρχονται. Υπάρχουν θέματα ανταγωνιστικότητας, υπάρχουν θέματα ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στην τοπική παραγωγή και τις εισαγωγές. Αυτό καθορίζεται από ποσοστώσεις δασμολογικές, καθορίζεται από το κόστος της εργασίας, από ειδικές συνθήκες σε διάφορες χώρες παραγωγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λειτουργούν τα συστήματα εις βάρος των προϊόντων μας και αυτό αφορά το σύνολο των εμπορικών συμφώνιων με τις τρίτες χώρες. Θεωρώ ότι πρέπει να τηρούμε πολύ αυστηρός ε, τους κανόνες και δεν θα θυσιάσουμε τα υγειονομικά μας μέτρα και τα φυτοϊγειονομικά μας μέτρα για περισσότερη ελευθερία. Τα φυτοϊγειονομικά μέτρα υπάρχουν, υπάρχουν ε, ως ε, προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και πιστεύω ότι θα πρέπει να τα τηρήσουμε. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι αυστηροί έλεγχοι για τις εισαγωγές, κυρίως για εισαγωγές υψηλού κινδύνου, όπως τα ζώντα ζώα και τηρούνται. Ε, το δικαστήριο δε ε, έλαβε προσφάτως μία απόφαση για τις εισαγωγές ε, και είχαμε και σχετική έκθεση. Η έκθεση είναι θετική για τους ελέγχους που κάνουμε και για το, όσα κάνουμε και στα σύνορα. Αλλά φυσικά υπάρχουν σχόλια και αυτό απαντά και στο ερώτημα που μου ετέθηκε για το τι θεωρώ εγώ για τους συνοριακούς ελέγχους και, και την εφαρμογή των ελέγχων. Σε γενικές γραμμές, σε θέματα ασφαλείας, είμαι θετικός. Θεωρώ ότι υπάρχουν αποτελέσματα και υπάρχουν καλά αποτελέσματα βάσει των ελέγχων μας στα σύνορα. Αυτό όμως που διαπιστώνουμε είναι ότι επειδή το σύστημα επιβλήθηκε τα τελευταία χρόνια με πολύ κατακαιρματισμένο τρόπο. Νομίζω έχουμε 12 διαφορετικούς κανονισμούς που ασχολούνται με το θέμα. υπάρχουν ε, πολλοί έλεγχοι που δεν είναι επικεντρωμένοι στα σωστά στοιχεία. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι Ε, ε, η διοίκηση που προωθούμε για τους ελέγχους είναι ανάλογη με αυτό που περιμένουμε ως αποτέλεσμα και αξιολογείται με βάση αυτά που επιθεωρούμε. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μία μεμονωμένη προσέγγιση ενιαία για όλες τις περιπτώσεις, γιατί νομίζω ότι αυτό θα ε, δημιουργήσει πρόβλημα στη δυνατότητα ελέγχου που έχουμε και τελικώς θα έχουμε μείωση των ελέγχων. Αν είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό που θέλουμε και βασιζόμαστε στον έλεγχο για τους κινδύνους, νομίζω ότι τελικώς θα έχουμε καλά αποτελέσματα και θα υπάρχει ποιοτικός έλεγχος. Όσον αφορά τώρα τις αξιολογήσεις στα σύνορα, υπάρχουν προγράμματα επιμόρφωσης ε, για τις ε, τελωνιακές υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Γνωρίζω ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά και εμείς δεν καθόμαστε στα αυγά μας, αλλά έχουμε ε, προγράμματα συνεχώς προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είναι λογικά τα επίπεδα αξιολόγησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσφάτως υιοθότησε και μία έκθεση για τους ελέγχους, ε, η οποία είναι πλέον στα χέρια του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βλέπουμε τι γίνεται με τις εισαγωγές. Επομένως, το Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η πολιτική μας για τις εισαγωγές. Οι διαπραγματεύσεις τώρα με τη Μερκοσούρ είναι ένα σημείο στο οποίο εμένουμε και εδώ ε, θα είμαι πολύ αυστηρός. Θέλουμε να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση ε, στις προδιαγραφές, ε, δεν θέλουμε να υπάρχει καμία ε, μείωση στις προδιαγραφές. Όσον αφορά τώρα το τι πιστεύουμε για τα ζωικά άλευρα, όπως είπε και ο κύριος Νίκολσον, περάσαμε μία πολύ προβληματική περίοδο, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε πολλές διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε ανάλογα φαινόμενα. Και χαιρόμαστε νομίζω γιατί θεωρούμε ότι η δράση μας απέδειξε στην πράξη ότι καταφέραμε να εκριζώσουμε τις νόσους και παρά το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα θέματα αυτά, θα πρέπει να αντιδρούμε ανάλογα με την κατάσταση. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε είναι τα ζωικά άλευρα από χείρους να χρησιμοποιούνται για ε, τροφές τα πολλορικά και ζωικά άλευρα από πουλορικά να χρησιμοποιούνται ε, ζωοτροφές χείρων. Αλλά τα ζωικά άλευρα μυρικαστικών να εξακολουθούν να απαγορεύονται. Φανταζόμαστε ότι θα έχουμε στοιχεία μέχρι το τέλος του 2011 για το τι ακριβώς θα γίνει με τα ζωικά άλευρα. Τώρα, για τις ε, ταυτότητες ε, των ε, εγωπροβάτων. Πήγα προσωπικώς ε, σε μια κτηνοτροφική μειονάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δω ε, ιδίως όμως τη διαδικασία για τις ταυτότητες των εγωπροβάτων. Διαπίστωσα τι επιπτώσεις υπάρχουν ο Γεωργός χρησιμοποιούσε ταυτότητες που δεν πληρούσαν απλώς και μόνο τις ζωικές μας απαιτήσεις, τις νομικές μας απαιτήσει, αλλά εφιώς το είχε επεκτείνει και στην καλή διαχείριση της κτηνοτροφικής του μονάδας. Και νομίζω ότι υπήρχε ένα μεγάλο άχθος για τη διαχείριση του θέματος και ίσως να οφειλόταν και στο γεγονός ότι υπήρχαν και επιπλέον λειτουργίες σε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Ε, η κτηνοτροφική μας υπηρεσία, ιατρική μας υπηρεσία πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σκοτία την περασμένη εβδομάδα. Εξετάζουμε λοιπόν την κατάσταση. Ε, γίνονται έλεγχοι επιτόπου και θα περιλάβουν και την Ιρλανδία και την Ισπανία και την Πορτογαλία και θα υπάρξει και μία έκθεση για τα διδάγματα που αντλήσαμε από αυτές τις ε, ελεγκτικές αποστολές ε, αργότερα εντός του 2011. Το θέμα των ταυτοτήτων αυτών είναι πολύ σημαντικό. Αναφέραμε και άλλα θέματα, αλλά όταν ασχολούμαι με τα διάφορα θέματα που αφορούν την υγεία των ζώων, υπάρχει η εξής αντίφαση στα όσα κάνουμε η κλωνοποίηση. Δεν θα ξεκινήσω εδώ τώρα τη συζήτηση για την κλωνοποίηση, θα τα πω αργότερα. Αλλά ένα από τα ε, θέματα που μας αφορά στην κλωνοποίηση είναι η χνηλασιμότητα. Όταν συζητάμε την χνηλασιμότητα, αυτό μας ενδιαφέρει, που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει χνηλασιμότητα. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε περισσότερες ε, ταυτότητες. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που μας λένε ότι θα πρέπει να αναλύσετε τι επιπλέον άχθος έχουμε όταν ε, ε, χρησιμοποιείτε ταυτότητες για άλλους λόγους στα εγωπρόβατα. Εδώ συζητάμε επίσης και την εισαγωγή νέων μέτρων τα οποία θα απαιτούν και πάλι ταυτότητες. Θα πρέπει λίγο να καταλάβουμε και πώς έχουν τα πράγματα. Τώρα, για τους κλωβούς ε, των τόκων ορνήθων. Ε, από ό,τι κατάλαβα, αυτή είναι βασική προτεραιότητα της Επιτροπής σας. Πόσο χρόνο έχω ρετάει ο Επίτροπος. Δυστυχώς δεν ακούμε την απάντηση. Για τους ε, κλωβούς, λοιπόν, το θέμα είναι σημαντικό. Μόλις ανέλαβα καθήκοντα, ήταν από τα πρώτα θέματα που χρειάστηκε να με απασχολήσουν. Δύο θέματα είναι σημαντικά εδώ. Καταρχάς, δεν θα επαναχωρήσουμε. Υπάρχει νομοθεσία συγκεκριμένη για τη θέση μας και το ανέφερα αυτό ρητό στο Συμβούλιο κατόπιν ετήσεω κάποιων κρατών μελών να αναβληθεί η ημερομηνία θέση ε, σε ισχύ τη νομοθεσία και αρνήθηκα δι. Και το έκανα αυτό διότι συμφωνώ με ένα από τα σχόλια που ακούσαμε εδώ, διακυβεύεται η αξιοπιστία μας επί του θέματος και θεωρώ ότι θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται αποδεκτό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κανόνε και μια συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο, αυτά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Και επειδή το έχω βιώσει και στη χώρα μου, κάποιοι ε, αρχίζουν να σκέφτονται ότι πρέπει να εφαρμόσουν κάτι όταν ε, μένει μόνο μια εβδομάδα για την εφαρμογή του. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο υπάρχουν οι μεταβατικέ περίοδοι. Θα πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδο για να βοηθήσουμε κάποιον να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Και θεωρώ ότι ήταν 12 χρόνια εδώ η μεταβατική περίοδο. Είχαμε 12 χρόνια να προσαρμοστούμε για τους ε, κλοβού και τι φωλιέ και νομίζω ότι αυτό ήταν επαρκέ χρονικό διάστημα για να συμμορφωθούν όλοι με τι προδιαγραφέ. Ωστόσο υπάρχουν χώρε που όπω είπατε κι εσεί δεν συμμορφούνται. Συζητούσα με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο επί του θέματο και επέμενα στο γεγονό ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον πληροφορίε. Εσεί μου ζητήσετε κάποιο εφευρωικό σχέδιο. Μπορεί να έχουμε πολλά εφεδρικά σχέδια το ένα πίσω από το άλλο, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το πώ έχει κατάσταση επιτόπου. Διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αρκετά στοιχεία. Ο τελευταίος αγορητής μας είπε ότι θα καταστρέψουμε τις όρνηθες. Ένας συναδέλφος μου είπε ότι οι Ιταλοί εχθές κατάσχεσαν ένα εκατομμύριο όρνηθες λόγω των κλοβών. Δεν ξέρω τι γίνεται τι θα τις κάνουν και ένα εκατομμύριο όρνηθες, αν όντω ισχύει ότι κατασχέθηκαν ένα εκατομμύριο όρνηθες. Για λόγους ε, ευημερίας των ζώων ελπίζω να μην ε, τις φάξουν, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο κύριος Αγνιού αναφέρθηκε πολύ καλά στις επιπτώσεις των αποφάσεων που, που θα λάβουμε. Ε, επιπτώσεις για τον ε, τομέα, για την αγορά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εισαγωγέ ε, αυγών στην Ευρώπη. υπάρχει επάρκεια. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Πραγματικά περιμένω να λάβω όλες τις πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε με ευφυή και αναλογικό τρόπο να εξετάσουμε τις επιπτώσεις όσων θα κάνουμε. Θα πρέπει να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς κανόνες. Δεν μπορούμε να έχουμε αυγά από μονάδες που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τους κανόνες και να θεωρούμε ότι αυτά θα είναι ανταγωνιστικά ε, με τα αυγά σε χώρες που έχουν συμμορφωθεί προς τους κανόνες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία οποιοδήποτε σχεδίου μας. Από εκεί και πέρα το τι μελιγενέστε θα εξαρτηθεί. Αν διαπιστώσω για παράδειγμα ότι η Πολωνία, παράδειγμα σας δίνω, και έχει 80% μη συμμόρφωση, τι θα κάνουμε. Θα καταστρέψουμε την αγορά της Πολωνίας και θα εισάγουμε αυγά από αλλού. Δεν σας τα λέω ως γεγονότα, σας δίνω απλώς παραδείγματα. Αλλά αυτά καταδεικνύουν ότι είναι σημαντικό να έχουμε όλα τα στοιχεία αναχείρα, ώστε αυτή τη στιγμή λάβουμε απόφαση και υπάρξει μια πρόταση, να είναι μια πρόταση που θα ε, είναι βιώσιμη και θα μπορούμε να την υπερασπιστούμε κιόλα. Αυτή τη στιγμή 15 χώρες δεν έχουν στείλει πληροφορίες. 15 χώρες. Από την τελευταία φορά που μίλησα στο Συμβούλιο μου είπαν ότι τέσσερι από τις χώρες αυτές έχουν ήδη στείλει πληροφορίε. Κάποιοι λένε ότι έχουμε πλήρη συμμόρφωση, απλώς δεν θα στείλαμε τις πληροφορίε. Ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς παρακολουθούμε συνεχώς ε, το ζήτημα και θέλουμε να λάβουμε τι πληροφορίε. Αυτή είναι η θέση μας για το ζήτημα αυτό. Τώρα για τις διοξίνες. Βρισκόμαστε σε επαφή με την γερμανική κυβέρνηση σε μόνιμη βάση από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Έχω μιλήσει τηλεφωνικά με τον Υπουργό επανειλημμένα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι το θέμα των διοξινών μας δείχνει τελικά ότι το σύστημά μας λειτουργεί. Αν το σύστημά μας ε, γίνει αντικείμενο σωστής διαχείρισης, λειτουργεί. Ανεξάρτητα από τις οδηγίες τις οποίες περνάμε, δεν έχουμε εγγυήσει ότι δεν θα υπάρξει κάποιος εγκληματίας ο οποίος θα προσπαθήσει να βάλει τρικλοποδιά στο σύστημα. Εμείς θα πρέπει να έχουμε σωστές πολιτικές και σωστές διαδικασίες έτσι ώστε αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε να προειδοποιούμε θα το ταχύτερο δυνατόν και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να αντιδράσουμε με μεγάλη ταχύτητα. Ο τρόπος ανείχνευσης που έχουμε του προβλήματος λειτουργεί και η Γερμανία το είδε αυτό, μπόρεσε να εντοπίσει του ε, τους τις αιστείες από τις οποίες προκλήθηκε το πρόβλημα προχώρησε στο να κλείσουν κάποιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να απαγορευτεί η επεξεργασία προϊόντων από τις φάρμες αυτές, από τις μονάδες αυτές. Και κατέληξαν στο ότι δεν υπήρχε τρομερός, ιδιαίτερος μάλλον κίνδυνος για τα τρόφιμα Φυσικά ε, υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν μέτρα ε, εναντίον των εταιριών οι οποίες κυκλοφόρησαν κάποιες ζωοτροφές οι οποίες ήταν μολυσμένες. Το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, με λίγα λόγια δούλεψε. Έχουμε κάποια συστήματα εν λειτουργία για τα οποία μερικές φορές παραπονιόμαστε βέβαια θεωρούμε ότι δημιουργούν επιπλέον κόστος, επιπλέον βάρη, αλλά αυτά τα προβλήματα νομίζω ότι αντιμετωπίζονται και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο χρήσιμα είναι. Με ρώτησε ο κύριος Χλώσιν, ο κύριος γιατί είμαι κατά της μεθόδου ανείχνευσης των συγκεκριμένων αυτών προϊόντων. The αυτό αυτός ο θετικός χαρακτήρας των ζωοτροφών θα πρέπει να καθορίζεται από την σωστή, ε, θα έλεγα, προσαρμογή τους και τη συμβατότητά τους με τους ισχύοντες κανόνες. Αν ένα τέτοιο προϊόν αναγνωρίζεται ότι πληρεί τους συγκεκριμένους κανόνες, δεν νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να διευκρινίζουμε ότι η ζωοτροφή αυτή είναι θετική, γιατί τότε ποια είναι η αρνητική. Νομίζω ότι ε, αυτό είναι το βασικό μου θα έλεγα επιχείρημα ε, ε, κατά της μετακίνησής μας προς την κατεύθυνση την οποία ανέφερε και ο Σχόσλινγκ. Για τα γενετικά τροποποιημένα τώρα, εμείς έχουμε ήδη κάνει τις προτάσεις μας και πράγματι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων. Εμείς ε, ε, εκλεπτύναμε αν θέλετε σε επίπεδο λεπτομέρειας τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τους λόγους και τα γιατί τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να βασίσουν τις απόψεις τους, τις αποφάσεις τους. Νομίζω ότι σιγά σιγά καταλήγουμε σε μια γενικότερη κατανόηση της κατάστασης και των λόγων που οδηγούν τα κράτη-μέλη να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να παίρνουν τις αποφάσεις. Θα έλεγα αυτό έχει σημασία. Εγώ αν ήμουν ένα κράτος μέλος, η δική μου χώρα, αν ήμουν υπεύθυνο στη δική μου χώρα, θα έλεγα ότι η χρήση της γης είναι ένα βασικό, θα έλεγα, μια βασική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, νομίζω ότι οι χώρες θα πρέπει να έχουν την εξουσία, την αρμοδιότητα να αποφασίζουν επί τη βάση οικονομικών και κοινωνικών λόγων θα έλεγα, αντικειμενικών στόχων, να κατανέμουν ε, και να, την γη και να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται ο καλλιεργητής στη γη. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς ότι μία χώρα θα είναι μία χώρα στην οποία θα καλλιεργούνται μόνο, θα έλεγε, οργανικές, οργανικές καλλιέργειες. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η χώρα, να πει ότι στους τομείς αυτούς θα υπάρχουν ε, οργανικές καλλιέργειες και σε κάποιους άλλους τομείς θα υπάρχουν ε, εντατικές καλλιέργειες. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα έλεγα με φυσικό τρόπο εναπόκειται στα κράτη-μέλη να το αποφασίζουν. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι όμως. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εάν η αδειοδότηση για την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων βασίζεται στο ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και δεν υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει ε, να, να αντιμετωπίζεται εκ νέου από τις διαδικασίες που ακολουθούν τα κράτη-μέλη για να καταλήγουν σε αποφάσεις. Σχετικά με αυτά που είπε ο κ. Μποβέ για τα γενετικά τροποποιημένα, ξέρετε τι προσπαθώ να κάνω στα γενετικά τροποποιημένα. Έχουμε τη λεγόμενη νέα διαδικασία, η οποία έχει προτεθεί από την ΕΦΣΑ, για την διαδικασία διοδότησης. Εγώ αυτήν την διαδικασία την έχω θέσει σε δημόσια διαβούλευση. Ήδη έχουμε οργανώσει δύο πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια με επιστήμονες και πολιτικούς από όλε τις πλευρές και από όλους τους τρόπους σκέψης. Έγιναν ελεύθερες συζητήσεις, όχι απλά να μεταφέρουν τις απόψεις τους, αλλά να ακούσουν και τις αντίθετες απόψεις. Το τι προσπαθώ να πετύχω μέσα από όλα αυτά είναι να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε ένα σύστημα στα πλαίσια του οποίου οι περισσότεροι από τους εμπλεκομένους, δυστυχώς όχι όλοι, θα συμφωνήσουν με τις διαδικασίες αδειοδότησης οι οποίες είναι σε ισχύ σε κάθε κράτος μέλος. Εγώ θέλω να έχουμε μια διαδικασία στη διάθεσή μας που να ικανοποιεί την πλειοψηφία των εμπλεκομένων και των γεωργών και των καταναλωτών και τους των επιστημόνων οι οποίοι να μπορούν να κάνουν τους δικούς τους ελέγχους, ανεξάρτητοι επιστήμονες που να παρακολουθούν τα, το τι συμβαίνει μετά τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Και πέραν αυτού εγώ και οι υπηρεσίες μου πάρα πολύ σύντομα, σε λίγες μέρες αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους για τις κοινωνικο-οικονομικές πλευρές της χρήσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Είναι μια ανάλυση του τι ακριβώς έχουμε συλλέξει από τα διάφορα κράτη-μέλη. Και ε, αυτά τα οποία μας έδωσαν τα κρατη δεν ήταν και πάρα πολλά πρέπει να ομολογήσω. Εκ των πραγμάτων τα στοιχεία που πήραμε δεν ήταν πλούσια, δεν ήταν στοιχεία θα έλεγα πραγματικής παρακολούθησης των, της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων γιατί περισσότερες χώρες έτσι κι αλλιώς δεν καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένα απλά παρουσίασαν το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Εμείς προσπαθήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά τα στοιχεία να τα και όπως είπα θα δημοσιεύσουμε την έκθεσή μας το ταχύτερο δυνατόν. Επιμένω ως προς αυτό γιατί τα γενετικά τροποποιημένα ε, εντάσσονται στα πλαίσια της λογικής της υπεύθυνης καινοτομίας θα έλεγα. Μιας καινοτομίας ευεργετικής για το σύνολο της κοινωνίας. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να δούμε είναι το τι πλεονέκτημα μπορούμε να βγάλουμε από κάθε προϊόν το οποίο προτείνεται στην αγορά. Εγώ έχω κάνει αυτές τις δηλώσεις, επαναλαμβάνω δεν είμαι υπέρ κατά των γενετικά τροποποιημένων, δεν είμαι υπέρ ή κατά της κλωνοποίησης, αλλά είμαι ανοιχτός στην καινοτομία. Και δεν θα ήθελα να κλείσουμε τον δρόμο στην καινοτομία, θα ήταν αρνητικό για τις κοινωνίες μας αν απαγορεύαμε την καινοτομία, θα ήταν αρνητικό για τον Ευρωπαίο πολίτη το να κλείσουμε τα αυτιά μας, να κλείσουμε τα μάτια μας και να αγνοήσουμε τις καινοτομίες οι οποίες υπάρχουν γύρω μας. Δεν είναι θέμα εμπορίου, δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είναι θέμα του μέλλοντός μας. Θα πρέπει να είμαστε δεκτικοί, ανοιχτοί, να είμαστε φυσικά ε, ε, προληπτικά έτοιμοι να αντιδράσουμε σε προβλήματα με μια κάποια αναλογικότητα και να έχουμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Εγώ τον τελευταίο χρόνο που είμαι εδώ και κάνω αυτή τη δουλειά σε εισαγωγικά είναι ότι μερικές φορές η επιστήμη είναι χρήσιμη ε, και την δεχόμαστε, αλλά όταν θεωρούμε ότι δεν μας δίνει τις απαντήσεις τις οποίες επιδιώκουμε, δεν την λαμβάνουμε υπόψη. Πρέπει να βασιζόμαστε λοιπόν στις επιστημονικές, ε, ε, στα επιστημονικά στοιχεία και για το θέμα των γενετικά τροποποιημένων ελπίζω να υπάρξει μια αντικειμενική κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή λέει ο Επίτροπος και να καταλήξουμε σε κάποιες θέσεις. Για την κλωνοποίηση τώρα, για μια ακόμη φορά όταν έκανα τη συνέντευξη τύπου με ρώτησαν θα φάτε κλωνοποιημένο κρέας και είπα βεβαίως και θα φάω κλωνοποιημένο κρέας γιατί θεωρώ ότι είναι ασφαλές. Το κλωνοποιημένο κρέας ε, δεν ε, υποστηρίζει κανείς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορεί να υπάρξει θέμα υγείας στην κατανάλωσή του. Αλλά όμως υπάρχουν θέματα που πρέπει να δούμε. Το βασικό πρόβλημα με την κλωνοποίηση είναι φυσικά το θέμα της ευημερία των ζώων. Δεν είναι θέμα υγείας και υγιεινής. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να τα δούμε τα πράγματα όπως πρέπει. Κάποιος άλλος με ρώτησε αν θα προστατεύσω τον καταναλωτή από ε, τα κλωνοποιημένα κρέατα. Δεν υπάρχει θέμα προστασίας, δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει έκθεση σε κίνδυνο. Παρόλα αυτά Έχουμε κάποιες αξίες όπως το θέμα της ευημερία των ζώων και εμείς εμένουμε στις αξίες αυτές, στις αρχές αυτές και η πρόταση που έκανα ήταν ε, ναι μένα η κλωνοποίηση είναι ένα πρόβλημα σε σχέση με την ευημερία των ζώων, υπάρχουν θέματα ως, ως προς αυτό, και γι' αυτό εμείς στείλαμε το μήνυμα στην Ευρώπη, μιλήσαμε για το moratorium για την ε, ε, διατροφή ε, με κλωνοποιημένα ζώα και με την απαγόρευση χρήσης τροφίμων από, που προέρχονται από κλωνοποίηση. Μου ζήτησαν να κάνω μια νομοθετική πρόταση και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα μέχρι το τέλος του 2013 σχετικά με την αντιμετώπιση συνολικότερα του θέματος αυτού. Εγώ δεν θέλω να πάρω ε, τέτοιου είδους θέσεις και δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους προτάσεις νομοθετικές σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Απαιτείται να έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία. Σήμερα δεν τα έχουμε τα στοιχεία αυτά. Υπάρχει μια πλήρως ελεύθερη κατάσταση με τα παράγωγα ζώα, με ε, τα ζώα που κληρονομούν το DNA, με τα κλωνοποιημένα ζώα. Πρέπει να υπάρξει κάποιος κανόνας, κάποια ρύθμιση γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει και εδώ τίθεται κυρίως το θέμα της ανιχνευσιμότητας του αναπαραγωγικού υλικού. Ε, πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το από πού προέρχεται. Να σας πω μια μικρή ιστορία. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέμα της κλωνοποίησης, μου έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθήσει κανείς να ανιχνεύει την προέλευση των ζώων των οργανισμών. Πράγματι είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι θέμα κανόνων, τεχνικά είναι δύσκολο να το κάνει κανείς αλλά όταν είπα πόσα ε, ζώντα ζώα εισάγουμε και μου είπαν 50 ζώα, αριθμός 50. Οπότε είπα πού είναι το πρόβλημα αν εισάγουμε μόνο 50 ζώα. Λοιπόν, πριν παίρνουμε κάποιες αποφάσεις πρέπει να έχουμε, πάρει τα, να έχουμε συλλέξει τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι ότι δεν εισάγουμε κλωνοποιημένα ζώα. Εάν λοιπόν πράγματι πρέπει στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και της ανιχνευσιμότητας της προέλευσης των ζώων και της καταγωγής των ζώων. Πιέζουμε το Συμβούλιο και προς την κατεύθυνση αυτή. Να υπάρξει ε, ε, επίσης ε, θέμα ετικετοποίησης βοήου κρέατος το οποίο προέρχεται από συγκεκριμένο αναπαραγωγικό υλικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει όταν έχουμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας μια μελέτη των επιπτώσεων. Όταν μιλάμε για ετικετοθεσία τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, φαντάζομαι χάμπουργκερς και αλαντικά και παγωτά ίσως, δεν ξέρω. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία μελέτη επιπτώσεων για να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες. Δεν υπάρχει θέμα κινδύνου υγείας. Το θέμα... Το θέμα των ακογόνων ας ζώων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, ρυθμιστεί μέσω της ετικετοθεσίας. Λοιπόν, αυτά είχα να πω σε σχέση με την κλωνοποίηση. Είναι κρίμα που η κλωνοποίηση χρησιμοποιήθηκε σαν μοχλός για τα καινοτόμα τρόφιμα, για την οδηγία για, να, για τα καινοτόμα τρόφιμα. Νομίζω ότι χάσαμε μια καλή ευκαιρία. Νομίζω ότι η οδηγία αυτή θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη βεβαιότητα και στους καταναλωτές και στους παραγωγούς. Εγώ ζήτησα από τις υπηρεσίες μου να κινηθούν γρήγορα και να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν, θα έλεγα, την, να επαναπροτείνουν την οδηγία για τα καινοτόμα τρόφιμα και εδώ όμως χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Δεν θα ήθελα εγώ σε καμία περίπτωση να φανεί ότι σας πιέζω γιατί έχω συμφέροντα ή όχι, όχι, εγώ σας ζητώ κάτι πολύ ξεκάθαρα δεν προωθώ τα καινοτόμα προϊόντα για συγκεκριμένους λόγους συμφέροντος. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται αυτή η οδηγία ή έχουμε μια οδηγία η οποία όμως όλοι συμφωνούμε ότι απαιτείται να αλλάξει και θα ήθελα αυτή η νομοθετική πρόταση για τα καινοτόμα τρόφιμα να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν υπάρξει αποφάσεις και για το θέμα της κλωνοποίησης θα πρέπει επίσης να κινηθούμε γρήγορα και να καταλήξουμε σε μια νομοθετική πρόταση ικανοποιητική. Αυτό θα ήθελα να δω να γίνεται. Αλλά θα ήθελα η διαδικασία να είναι διάφανη, η συζήτηση να είναι διάφανη και με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Θέλω να κάνω λοιπόν συζητήσεις μαζί σας πριν κάνω προτάσεις. Αυτά. Να κάνω μια διόρθωση για τα αυγά που προέρχονται από τόκες ε, ε, όρνηθες. Περιμένουμε τα στοιχεία για τα αυγά από τα κράτη-μέλη. Αυτά. Λοιπόν για την κλωνοποίηση και τα καινοτόμα τρόφιμα δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα το οποίο δεν κάλυψα. Ίσως να υπάρχει συγγνώμη. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ το Τζον Ντάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ διότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Σαφώς βέβαια υπάρχει ακόμα διχογνωμία, υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες σε κάποια θέματα, αλλά νομίζω ότι η επιστημονική προσέγγιση που χρησιμοποίησατε, που δεν ήταν καθόλου ιδεολογική, θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε αυτή την τόσο ευαίσθητη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό διακοπή και θα συνεχίσουμε με το σημείο υπαριθμών 11, την έκθεση Μάρτιν ε, Χόσλινγκ. Ένα λεπτάκι, μην κουνηθεί κανείς.